μεσημέρι και τη, η επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ, προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφή, προκλήσει και ευκαιρίε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρώτο ομιλητή, ο ίδιο ο εισηγητή, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο ΟΗΕ έχει συγκαλέσει για την επόμενη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη τέτοια παγκόσμια διάσκεψη για τα θέματα αυτά. Στο δρόμο λοιπόν για την Κωνσταντινούπολη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε μια ανακοίνωση που κρίνει πολύ θετικά η δική μου έκθεση και που παρακολουθεί όλα τα θέματα αυτά. Αύριο θα ψηφίσουμε και το Συμβούλιο έχει προετοιμάσει και κάποια συμπεράσματα σχετικά τα οποία σίγουρα του χρόνου, πιο κοντά στη χρονική στιγμή της διάσκεψης, θα λάβουν την οριστική τους μορφή. Η έκθεσή μου προσπαθεί να δώσει μια απόκριση σε τρία θέματα. Καταρχήν, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια τέτοιου είδους ανθρωπιστική διάσκεψη αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, ποιοι είναι οι στόχοι του οποίου θέλουμε να πετύχουμε στην Κωνσταντινούπολη. Και τρίτον, τι ρόλο θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Για να απαντήσω στην πρώτη μου ερώτηση, δεν είναι πως χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια διάσκεψη, γιατί εδώ και 25 χρόνια εγκρίθηκε το Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Σύστημα και με την πάροδο του χρόνου χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πιο βαθιοί λόγοι. Έχει αλλάξει δραστικά ο κόσμος γύρω μας μέσα στα τελευταία 25 χρόνια και το ανθρωπιστικό σύστημα που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να αποκριθεί στις νέες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αντιμετωπίζουμε ανθρωπιστικές κρίσεις πιο δύσκολες, πιο σοβαρές, πιο πολλές από ό,τι ποτέ και σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Έχουμε παράλληλα μεγαλύτερες κρίσεις που προκαλούν φυσικές καταστροφές όπως επίσης και πολεμικές σειράξεις. Και έχουμε λιγότερα μέσα στη διάθεσή μας για να δώσουμε μια απάντηση σε αυτές τις κρίσεις οι οποίες διαρκούν περισσότερο γιατί πολλές φορές διαρκούν και 30 χρόνια. Ε, είναι δηλαδή αγκυλώσεις ουσιαστικά, τις οποίες δυσκολευόμαστε να ξεπεράσουμε. Ποιες είναι οι επιπτώσεις. Μεγαλύτερους αριθμούς προσφυγών από ό,τι ποτέ. 40 εκατομμύρια περίπου για το 2015. Και το ίμιση είναι παιδιά, ένα μεγαλύτερο κομμάτι ανθρώπων που χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. 100 εκατομμύρια άτομα περίπου πέρυσι. Αν τους βάλουμε όλους αυτούς μαζί, θα ήταν η δωδέκατη σε πληθυσμό χώρα του κόσμου. Για να σας περιγράψω περίπου γιατί μέγεθος μιλάμε θα ήταν η Γαλλία και η Ισπανία μαζί που θα χρειαζόταν ανθρωπιστική βοήθεια. Και έχουμε λιγότερα οικονομικά μέσα. Γιατί το 2015 χρειάστηκε ο ΙΕ να σταματήσει την παροχή κάποιας ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάποια σημεία του πλανήτη που επιγόντως χρειάζονται τη βοήθεια αυτή. Για να απαντήσω στη δεύτερη μου ερώτηση που ήταν τι θέλουμε να πετύχουμε στην Κωνσταντινούπολη, η έκθεσή μου έλαβε υπόψη την διαδικασία της παγκόσμιας διαβούλευσης που ξεκίνησε σε διάφορα σημεία του κόσμου και όπου συγκέντρωσε προτάσεις από διάφορους κλάδους οι οποίοι έχουν συστρατευθεί για να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε τέσσερις πυλώνες λοιπόν στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε. Πρώτα απ' όλα, παγκόσμια συνένεση για δράση η οποία θα επιβεβαιώσει τις αρχές, τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και το βασικό στοιχείο αυτής είναι η προστασία των ανθρώπων. Η συνένεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης πενταετές τουλάχιστον για να εφαρμόσουμε τα όσα θα αποφασίσουμε στη διάσκεψη. Δεύτερον, ένας κώδικας συμπεριφοράς που θα έχουμε συντάξει όλοι μαζί, όλοι οι δωρητές, όλοι οι συμμετέχοντες, χωρίς να ακολουθούμε κάποιες δυτικές επιταγές οπωσδήποτε, λαμβάνοντας υπόψη τους παγκόσμιους νόμους και τις θεμελιώδεις αξίες για την προστασία του ανθρώπου, έτσι ώστε τα συμπεράσματα της διάσκεψης να εφαρμοστούν στην πράξη. Τρίτον, θέλουμε ένα παγκόσμιο ταμείο ανθρωπιστικής βοήθειας για να προβλέπουμε, να είμαστε ευέλικτοι λειτουργικά και να είμαστε ασφαλείς λαμβάνοντας κάποιες ετήσιες ε, συνεισφορές. Γιατί μέχρι τώρα το σύστημα αυτό βασίστηκε σε εθελοντικές συνεισφορές. Θα πρέπει αυτές πια να είναι υποχρεωτικές. Τέταρτον, θα πρέπει να στηρίξουμε την προετοιμασία και την απόκριση η οποία θα δίδεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μία έκκληση λοιπόν πρέπει να απευθύνουμε έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η βοήθεια, να συμμετέχει και ο ιδιωτικό κλάδο όταν μπορεί να προσφέρει, γιατί έχει την εμπειρία, και ακολουθώντα τι ανθρωπιστικέ ε, ανάγκε που έχουμε για να προστατεύσουμε ανθρώπους. Το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα προσωρινά ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τη διάσκεψη αυτή να είναι επιτυχημένη και στη φάση της προετοιμασίας αλλά και στην μέγιστη εκπροσώπηση που θα έχουμε στην Κωνσταντινούπολη. Όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, διπλωματικά, ανθρωπιστικά, θα πρέπει να τα διαθέσουμε για να πετύχουμε αυτό το όρομα το οποίο θα προωθήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και που θα αλλάξουν σε βάθος την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα άτομα, τις ζωές τους, να εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια που είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε να πετύχουμε και εμείς οι ίδιοι να είμαστε αξιοπρεπείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο. Εκ μέρους της Επιτροπής, ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης και θα σας παρακαλέσω να περιορίσετε στα τρία σας λεπτά ή δυνατόν. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συναδελφοί. Ο ανθρώπινος πόνος έχει φτάσει επίπεδα που δεν έχουμε δει ποτέ πριν. Όπως είπε και ο κύριος Κεραίρο, πάνω από 100 ε, εκατομμύρια εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια, 60 εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και αυτά τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η επίκαιρη πρωτοβουλία. Η ανθρωπιστική βοήθεια να μπει στο επίκεντρο τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων και να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται η βοήθεια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικέ κρίσει. Αυτή η μεγάλη λοιπόν διάσκεψη κορυφή θα πρέπει να δώσει αποτελεσματικέ απαντήσει για την υλοποίηση τη ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να φροντίσει όντω να φτάνει στα χέρια των δικαιούχων αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Ιδιαίτερα λοιπόν πρέπει να φωτιστεί η όλο και εντυνόμενες, να παραβίαση, όλο και εντυνόμενες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη των πολιτικών σε αυτή τη συνοδοκορυφής. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο οι αρμόδιοι για τα ανθρωπιστικά να επιτύχουν τις λύσεις για τα κείμενα προβλήματα. Δεν μπορούν οι υπεύθυνοι για τα ανθρωπιστικά, ούτε και οφείλουν να ε, σηκώσουν όλο το βάρος μόνοι τους. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα είναι μόνο βραχυπρόθεσμη λύση και δεν μπορεί ούτε να αποτρέψει να περατώσει πολέμους ή ένοπλες συγκρούσεις. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, να γεννήσει οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Και αυτό με την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας, τη Συριακή, το βλέπουμε ξεκάθαρα όσο δεν εξευρίσκεται μια πολιτική λύση, όσο οι Σύριοι δεν μπορούν να έχουν κοινωνικές ευκαιρίες, η ανθρωπιστική μας βοήθεια προς τη Συρία και τις όμορες της χώρες θα είναι πάντα ανεπαρκής το γεγονός ότι αυτή η σύνοδο Κορυφή λαμβάνει χώρα στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας έχει τη δική της μεγάλη σημασία. Το δικό της συμβολισμό έχει αυτή η πόλη γιατί είναι το σημείο στο οποίο συνενώνονται χώρες ήπειροι πολιτισμοί και πρέπει να αποτελέσει ένα σύμβολο τη γέφυρα της οικονομικής και κοινωνικής προόδου και του σεβασμού στο περιβάλλον, ώστε να προστατευτούν καλύτερα, να υπηρετηθούν καλύτερα οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις. Πρέπει να προσφέρουμε δυνατότητα για συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα και γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι ηγέτες να ε, δείξουν διάθεση για συγκεκριμένες και σαφείς δεσμεύσεις στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο στην Κωνσταντινούπολη στην έξι μήνες θα έχουν κρίσιμη σημασία ώστε η Σύνοδος να ανέλθει στο ύψος των περιστάσεων, όπως οφείλει. Δική μου δέσμευση είναι με εταίρους σε όλο τον κόσμο να κάνω προσπάθειες για συνεννόηση εν ώψη τη Συνόδου. Το ίδιο πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερο έχει να διαδραματίσει ρόλο σε αυτό. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τους, ε, τις προσπάθειες, των ενδιαφέρον και την ανάμειξη στη συζήτηση για τη Σύνοδο αυτή των βουλευτών, ιδιαίτερα τον κύριο Γκερέρο Σαλόμ για την ε, δική του ηγετική πρωτοβουλία και ιδιαίτερα για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα αρχίσει να συζητείται αμέσως. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τη θέση της και την κοινοποίηση με την ανακοίνωση τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΔΕ Κοινοβούλιο θα πρέπει να ολοκληρώσει με την έγκριση της εκθέσεως αυτής τη δική του συμβολή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύνοδο. Και έτσι θα έχουμε μια ένα συλλογικό όραμα για το τι μπορεί να είναι μια αποτελεσματική, μια επιτυχημένη παγκόσμια σύνοδος κορυφής για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα μήνυμα σαφές προς όλους τους εταίρους μας ανά τον κόσμο και για την μεγάλη κρίση του προσφυγικού, όπου η Ευρώπη έχει αναλάβει το δικό της μεγάλο μερίδιο της ευθύνης με την πρωτοβουλία του Προέδρου Γιουνκέρ και της Επιτροπής που δείχνει ξεκάθαρα ότι η κρίση αυτή είναι μείζον προτεραιότητα για μας και ότι εδώ διακυβεύονται οι κύριες αρχές και αξίες της ανθρωπότητας και της αλληλεγγύης. Και αυτό θα επιδείξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη αναλαμβάνει λοιπόν το δικό της μερίδιο ευθύνη με τρεις κυρίως τρόπους. Πρώτα απ' όλα προσφέροντας υποστήριξη αρρωγή στους πρόσφυγες οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτοί. Δεύτερον, με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, δύσκολο όντως. Και τρίτον, με μια ε, συνολική αντιμετώπιση του συριακού προβλήματος και της κρίσης. Κάνουμε λοιπόν όπως είπα ό,τι οφείλουμε στο δικό μας μερίδιο της ευθύνης και έτσι ενισχύουμε και τη δική μας αξιοπιστία και γινόμαστε οι κύριοι συνήγοροι για να αναπτυχθεί αυτή η παγκόσμια ανταπόκριση, η παγκόσμια αντίδραση που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, λέει Πρόεδρο. Και τώρα ο κύριο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, εκ μέρου τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες των τεράστιων προκλήσεων αυτού του αιώνα. Ζούμε σε έναν πιο πλούσιο κόσμο, ο οποίος όμως είναι πιο εύθραυστος και όπου οι πολίτες είναι πιο ευάλωτοι. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις σημαίνουν, σημαίνουν ακριβώς ότι οι λαοί υποφέρουν και ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα μεταξύ των θυμάτων, ιδιαίτερα στις ένοπλες σειράξεις γιατί υφίστανται τη βία, τους βιασμούς και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη και να έχουν πρόσβαση για την αναπαραγωγική και σεξουαλική τους υγεία. Ελπίζουμε πραγματικά ότι η διεθνής διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για να ορίσουμε ένα νέο ανθρωπιστικό σύστημα για να ανταποκριθούμε στις αλλαγές. Ευχαριστώ κυρία Άννα Χέτ, Επιτροπή Γυναικών Ισότητας των Φύλων. Som rapportör för femutskottets yttrande så vill jag börja med που έχει σημασία να είναι να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που εργάστηκαν για την γνωμοδότηση στην Επιτροπή των Γυναικών. Έχουμε να κάνουμε με μία πολύ εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση για να βελτιώσουμε την εργασία μας στον ανθρωπιστικό τομέα. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση και νομίζω ότι ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ ε, είχε απόλυτο δίκιο όταν μίλησε για το ρόλο της ύπατης αρμοστίας ε, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά δεν έχουν τη σωστή ε, αντιμετώπιση ως προς την υγεία τους, την αναπαραγωγική υγεία και τη σεξουαλική υγεία. Θα πρέπει να προνοηθούν τέτοιες υπηρεσίες οι γυναίκες και τα παιδιά που ε, δυστυχώς υφίστανται αυτή τη βία δεν θα πρέπει να ε, τιμωρούνται διπλά επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή τη βία. Τώρα περνούμε στους ομιλητές εκ των ομάδων. Με την κυρία Ζαμπόρσκα πρώτη εκ του Ευρωπαϊκού Λυκού Κόμματος ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο για ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ ισορροπημένο και το οποίο νομίζω θα στηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες με κάποιες μικρές επιφυλάξεις. Ε, φέτος η Ευρώπη χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις μια ανθρωπιστικής κρίσης και μιας κρίσης προσφυγικής. Όλοι ξαφνιαστήκαμε από μια πραγματικότητα όπου εκατομμύρια διωγμένοι και διωκόμενοι μας χτύπησαν την πόρτα και μας δόθηκε μια ευκαιρία μέσω αυτής της άξαχνης έκπληξης να βρούμε καινούριου τρόπους για να διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους κρίσεις, για να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους κρίσεις και για να αντιδρούμε με πιο ταχύ τρόπο. Η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει πολύ επικοδομητικές προτάσεις που εξυπηρετούν αυτό το στόχο και με πολλή προσδοκία αντιμετωπίζω αυτή την διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης. Απογοητεύομαι βέβαια που δεν ήμασταν σε θέση να συμφωνήσουμε για το θέμα των αμβλώσεων ή για τις υποχρεωτικές συνεισφορές, θέματα τα οποία ακόμα είναι προτάσεις ε, στο χαρτί. Νομίζω ότι θα πρέπει η έκθεση αυτή να εγκριθεί με ευρύτερη συνένεση. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριο Νόιζερ για μισή λεπτό επίση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Ενρίκε. Η COP21 των Παρισίων ήταν μια μεγάλη διεθνής επιτυχία. Το... Τη μεγάλη αυτή ορμή, την παγκόσμια ορμή, χρειαζόμαστε και στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύω. Πρέπει να στεφθεί με επιτυχία η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το στηρίξει και με τη στάση της Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλήξουμε σε ένα καλό παγκόσμιο αποτέλεσμα. Οι ανάγκες και η κατεπίγουσα κυρίως ανάγκη δράσεως είναι πιο ορατή από ό,τι ποτέ. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα ζητήματα τα οποία παρισφρίουν, αλλά είναι δευτερεύοντα, δευτερεύοντα σημασία. Το κέρια σημασία είναι το θέμα των ανθρώπινων ζωών που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα εκατομμύριο Σύριοι στην Ευρώπη είναι σχετικά μικρό νούμερο. Γιατί από αυτού έχουμε το 1 τρίτο να είναι νέοι και παιδιά. Αδύναμα, δεν μπορούν να προστατευτούν μόνα του. Χρειάζονται τροφή, φάρμακα, στέγη. Και αυτό ισχύει και για τους 60 εκατομμύρια εκτοπιστέντες. Αριθμό ρεκόρ για περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε τρία χρόνια, μέσα στα 13 χρόνια από το 2002 στο 2015 έχουμε φτάσει στον αριθμό αυτό των εκτοπιστέντων. Και ελπίζουμε με την Κωνσταντινούπολη να εξασφαλίσουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ενρίκε, ευχαριστώ για την έκθεση. Αποτελεί πολύ καλή βάση για τις πραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ECR, ο κύριος Γκέρικε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανίδη, αγαπητέ Επίτροπε. Πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η Σύνοδος ε, του COP21 στο Παρίσι και με μεγάλους πανηγυρισμούς ο κύριος Φαμπιούς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση με επιτυχία της διασκέψεως. Εμείς ως Ευρωπαίοι, ε, εάν ε, προχωρήσουμε και πιέσουμε για μια μεγάλη ανθρωπιστική σύνοδο ε, μπορούμε να επιτύχουμε εξίσου καλά αποτελέσματα. Είναι μεγάλες οι κρίσεις, οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις, οι φυσικές καταστροφές. Ε, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο κόσμος μας χρειάζεται μια νέα κουλτούρα κάριτας, μια νέα κουλτούρα της αγάπης του πλησίων, δηλαδή του ελέους. Και σε αυτό νομίζω ότι μια μεγάλη σύνοδος δεν αρκεί μόνο, χρειάζονται μεγάλες και μεγαλειώδεις ιδέες. Την προηγούμενη εβδομάδα εκφράστηκαν προτάσεις για ένα μεγάλο φόρο, για ένα μεγάλο νόμο που θα φορολογούσε ε, υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας υπέρ των πιο φτωχών. Θα πρέπει να είμαστε θέσει να αντιδρούμε ταχύτερα στις ανθρωπιστικές καταστροφές. Πρέπει λοιπόν να η Πρόεδρος διακόπτη. Κύριε και ξεπεράσατε το χρόνο σας και δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω. Ευχαριστώ και η επόμενη ομιλήτρια εκ μέρους των Φιλελευθέρων, η κυρία Μπετσέρα Μπαστερετσέα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πίτροπε. Ζούμε σε μια κοινωνία επίγουσας ανάγκης και θα πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι. Δεν μπορούμε να παραμένουμε ακίνητοι. Αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ανάπτυξη Μα ε, μας οδηγούν στο να λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτή λοιπόν η διάσκεψη θα πρέπει να τιμηθεί στο υψηλότερο επίπεδο με παρουσίες ε, σε ε, επίπεδο αρχηγών κρατών όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από παντού. Κωνσταντινούπολη, ένα μέρος γεμάτο συμβολισμούς, ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους πρόσφυγες που συνοστίζονται στα σύνορα της Ευρώπης. Να δούμε πώς η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως όπλο πολιτικής και διπλωματίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται πια στον κόσμο. Είμαστε μεγαλύτεροι διορητές και θα πρέπει στη διάσκεψη αυτή να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα έτσι ώστε οι βασικές ανθρωπιστικές αρχές να γίνουν ε, σεβαστές όχι ατιμορρησία, προστασία για τις γυναίκες, το διεθνές νομικό πλαίσιο. Μην ξεχνάμε πως τα κράτη-μέλη δεν σέβονται πολλές φορές την διεθνή ε, νομή τάξη. Άρα λοιπόν πώς μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια συνεχή διάβρωση της προστασίας σε διεθνές επίπεδο και οι άμαχοι, οι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ που μετακινούνται στο εξωτερικό χρειάζονται όλο και περισσότερη προστασία από εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη και έχει έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και να προστατεύουμε όσους κινδυνεύουν. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουμε περισσότερη συνένεση σε διεθνές επίπεδο με ανθρωπιστική βοήθεια που θα λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα και που θα χρησιμοποιεί όσα μέσα διαθέτει. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Σάντσες ε, Καλντεντέι από την ε, Γοέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. 250 εκατομμύρια άτομα σήμερα επηρεάζονται από διάφορες ανθρωπιστικές κρίσεις. Πιο πολύ από ό,τι ποτέ χρειαζόμαστε μια ενορμανισμένη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν αξιολογούμε πολύ θετικά τα όσα έκανε ο κύριος Γκερέρο με την έκθεσή του και θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να επέμβουμε στη ρίζα του προβλήματος για την οικονομική ανισότητα μεταξύ ατόμων και μεταξύ κρατών. Είναι θεμελιώδες να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων, το δικαίωμα της ε, γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Χρειαζόμαστε μια δημόσια πολιτική η οποία θα είναι στεναρή στα θέματα αυτά και δεν θα ακολουθεί την λογική της ιδιωτικοποίηση όπως έχουμε στην έκθεση και για το λόγο αυτό θα δηλώσουμε άλλωστε και αποχή στην ψηφοφορία. Ναι, ο ιδιωτικό κλάδος, αλλά να εξυπηρετεί τους δικούς μας στόχους, τις δικές μας αξίες και να είναι υπεύθυνο και για τα όσα κάνει. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, είναι σημαντικό όλες οι πολιτικές μας να είναι συνεκτικές με τους στόχους που έχουμε, τους αναπτυξιακούς. Τι λείπει από αυτή την έκθεση αναφορές στο διεθνές εμπόριο, στην ευθύνη την εταιρική και στη, στο ευρωπαϊκό ε, εμπόριο όπλων. Δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε οποιαδήποτε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αστάθεια και οι κρίσεις και δεν δίνουμε λύσεις στις περιπτώσεις αυτές. Ευχαριστώ. επόμενη κυρία Χάουταλα, λεπτό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ετοιμαζόμαστε για την πρώτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τα ανθρωπιστικά σε μια περίοδο που απειλείται σοβαρά το ανθρωπιστικό δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αν σκεφτούμε όλες τις επιθέσεις σε μη πολεμικές ε, μονάδες, νοσοκομεία, σχολεία στο Αφγανιστάν, αυτά που ήδη υποφέρουν τόσο πολύ από τους πολέμους και τις αναπλές συγκρούσεις το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απειλείται και για άλλο λόγο και δυστυχώς και μέσα στο Κοινοβούλιο έχουμε πρόβλημα. Η εξέλιξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου δείχνει πλέον ξεκάθαρα τη χρήση του βιασμού συστηματικά ως όπλου σε ένοπλε συγκρούσει και πολέμους. Οι γυναίκες και τα κορίτσια που πέφτουν θύματα βιασμού έχουν αναπαλωτρίωτο και απερίφραστο δικαίωμα για άμβλωση ανεξαρτήτως της εθνικής νομοθεσίας τους μόνο και μόνο επειδή έχουν πέσει θύματα βιασμού σε συνθήκες πολέμου και σύγκρουσης. Πρέπει αυτό να το αποτρέψουμε. Πρέπει να ζητήσουμε να εξασφαλίζεται ασφαλής ε, άμβλωση σε τέτοιες περιστάσεις. Αυτοί που αρνούνται το δικαίωμα σε γυναίκες και τα κορίτσια αυτά απλώς είναι απάνθρωποι πιστεύω. Πρέπει αύριο να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην ιδέα για τη θέσπιση ενός διεθνούς ταμείου, ενός νέου διεθνούς Ταμείου, για το οποίο όμως δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή δεσμευτική συμμετοχή, γιατί δεν το βρίσκω τόσο λαμπρή ιδέα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής εκ μέρους ε, τη ε, Ομάδα Ευρώπη των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών, κύριος Κοράου. Χωρί μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια ε, ακολουθεί τα ίχνη άλλων διασκέψεων όπως της COP21, όπως της Νέας Υόρκης ή της Αντισαμπέμπα για την ανάπτυξη. Θα φτάσουμε σε μία θέση η οποία θα είναι αρκετά ισχυρή. Νομίζω ότι η εργασία του εισηγητή του κ. Ρωσαλόμ είναι μια πολύ καλή εργασία διαμεσολάβησης όπως ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υποστηρίξουμε την έκθεση. Βεβαίως η καλή εργασία αφορά και συμβουλές των ΜΚΟ που ασχολούνται με τέτοιες κατεπίγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να τη συγχαρούμε και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε όποιον δουλεύει επιτόπου για να μην γίνονται επιθέσεις σε ε, νοσοκομεία όπως των γιατρών χωρίς σύνορα. Η κυρία Μιρέιντονάνου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτή, αυτό το σχέδιο ανθρωπιστικής διάρθρωσης είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Θα πρέπει όμως να υπάρχει διαφάνεια και συντονισμός έτσι ε, ώστε να λάβουμε υπόψη ότι όλα αυτά δεν μπορούν να προωθηθούν ε, ως διατάγματα. Πολλοί έχουν πληγεί από τον πόμενο. Θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα το ανθρωπιστικό δίκαιο με τις επιτόπιες οργανώσεις. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και δεν εμπεριέχονται σε αυτό το σχέδιο ως προς την υποδοχή των προσφύγων ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μία παρηγορητική αγωγή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς που ασφικτιούν ολόκληρες οικογένειες μετατοπίζονται και υφίστανται τη βία καθημερινά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σοβαρά, διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσω να δεχτώ ε, την πολλωστή παγκόσμια διάσκεψη που δεν οδηγεί σε τίποτα. Ε, ο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα οποία προανέφερε, προανέφερθηκαν σε αυτό το στην από τον Πάπα Φραγκίσκο του, το δεύτερο ο, μας οδήγησαν να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και ο πόλεμος. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε την πλάτη στα θύματα. Η έκθεση του κυρίου Γκερέρο ανταποκρίνεται σε κάτι τέτοιο και αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια πραγματική δύναμη στον ανθρωπιστικό τομέα. Θα πρέπει να τηρήσουμε το μήνυμα του Παπα Φραγκίσκου γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θέματα βίας και βιασμών. Θα πρέπει να δεχτούμε όλους τους όρους του μήνυματος. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκερέρο για τις εξαιρετικές προτάσεις και το γεγονός ότι είναι ανοιχτός σε όλα τα μέτωπα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Φρανσίσκο Ασής. Αγαπητοί συνάδελφοι, το φιλοσοφικό μας υπόβαθρο μας οδηγεί στο να φέρουμε ευθύνη σε ένα τέτοιο ευμέγεθες ε, ε, πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και θα συνεισφέρουν έτσι ώστε η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης να είναι ένα πρόγραμμα δράσης που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού και να συνδέεται και με άλλα έγγραφα τα οποία τίθενται σε εφαρμογή όπως η ατζέντα η αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 και η ατζέντα της COP21. Θα πρέπει επίσης η ανθρωπιστική βοήθεια να λαμβάνει υπόψη την αρχή της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, καθώς και του ανθρωπισμού μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων αυτής της διάσκεψης, όπως προτείνεται από την έκθεση αυτή που ήταν πραγματικά εξαιρετική. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριος Νέιθαν Γκίλ. Ιρωνικό, Έτσι είναι. Που στην ε, Τουρκία γίνεται αυτή η μεγάλη σύνοδος. Όταν το Human Rights Watch καταγράφει με πολλαπλούς τρόπους την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από την Τουρκία, παρεμβάσεις στην πρόσβαση στο ίντερνετ, ε, περιστολή του δικαιώματος στην έκφραση, κλίματα κατά του τύπου και Βλέπουμε ότι ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την πρόσβαση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις παραβιάσεις αυτές. Όταν είμαστε υποτίθεται ένας θεσμός ο οποίος ε, ενστερνίζεται τις ανθρωπιστικές αξίες είναι τουλάχιστον παράδοξο αυτό. Μέρος, ε, μέλος του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία ταυτόχρονα αλλά απειλεί κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Και Είμαστε αφελείς αν νομίζουμε ότι μπορεί το εμπόριο, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει μια νοοτροπία αιώνων. Πρέπει να αποστείλουμε μήνυμα στον τουρκικό λαό ότι πρέπει να εκλέξει δημοκρατική κυβέρνηση και να προωθήσει θεσμούς και μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Γκίλ, ξεπεράστε το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος και διακόπτη. Ο κύριος Μωρίς Πόγκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Γκέρα Σαλόμ για την ε, δουλειά του στην έκθεση αυτή και προσωπικώ υποστηρίζω την έκθεσή του. Όπω αναφέρθηκε, η πρώτη ανθρωπιστική σύνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη στι 23 και 24 Μαου του 2016 στην Τουρκία και θα αποτελέσει ελπίζω ευκαιρία να δοθεί καλύτερη απάντηση στις καταστροφές, στις ανθρωπιστικές καταστροφές που είναι όλο και πιο πυκνές και συχνές. 200 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από ανθρωπιστικές καταστροφές, τεράστιες οικονομικές ανάγκες. Μέχρι το 2015 είχαμε τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανάγκες για ανθρωπιστική υποστήριξη. Ποσό ρεκόρ και για την ιστορία των Ηνωμένων Εθνών λοιπόν και θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις για να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπων. Η απάντηση θα πρέπει να είναι παγκόσμιου η ανσεμβελης Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ρόλο να δερματίσει ως κύριος και πρωταρχικός χορηγός. Πρέπει να παρέμβει και στην ανθρωπιστική βοήθεια και στη χρηματοδότηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των κρίσεων, ταυτόχρονα ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Βάιντενχολτσερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, συστηματική του δουλειά στην έκθεση και ελπίζω αυτή η σύνοδος να καταγραφεί ως επιτυχία όπως άλλωστε οφείλει. Η προσφυγική κρίση δείχνει πόσο κατεπίγουσα είναι η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις πού καταλήγουμε εάν δεν διατίθενται επαρκή μέσα, εάν δεν τηρούνται οι υποσχέσεις. Η κυρία Μέρκελ το Σεπτέμβριο στη Συνόδο για τους πρόσφυγες είχε πει τα εξής. Δεν προβλέψαμε ότι δεν θα αρκούσαν τα διεθνή προγράμματα με τη χρηματοδότησή τους και ότι θα πέθαναν από την πείνα οι άνθρωποι. Βεβαίως καλό είναι να βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά πρέπει να αλλάζουμε και στάση. Δεν έχουμε φτάσει όμως στο σημείο αυτό δυστυχώς. Γίνεται προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Συρία. Εμείς ως βουλευτές έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας. Τα κράτη-μέλη όμως ακόμη δυστυχώς διστάζουν και δεν τηρούν τα επισχημένα. Γι' αυτό χρειάζεται και ένας υποχρεωτικός μηχανισμός. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην εκούσια μόνο συμμετοχή. Και η ανάληψη ευθύνης ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέντα πριν από τη διαδικασία ευχαριστώ. είναι ο τελευταίος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με τα συγχαρητήρια προς τον ε, συντάκτη της έκθεσης που είναι εξαιρετική και νομίζω πως η διάσκεψη ήταν το σωστό βήμα για να ανταλλάξουμε απόψεις για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η κατάσταση Συρία, οι σειράξεις, η κλιματική αλλαγή είναι λίγες από τις κρίσεις με τις οποίες χρειάζεται να ασχοληθεί η διεθνής κοινότητα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποδοτική η ανθρωπιστική βοήθεια, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των όσων εργάζονται στον ανθρωπιστικό κλάδο, ξέρετε πως πάνω από 300 έχουν απαχθεί, σκοτωθεί ή τραυματιστεί το 2014. Η διεθνής αυτή διάσκεψη θα πρέπει να δώσει μια πολιτική όθηση έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η βοήθεια που θα προσφέρουμε και να εξασφαλίσει πως η βοήθεια αυτή θα κάνει πολλές κοινότητες και χώρες πιο σταθερές. Ευχαριστώ. Τώρα η διαδικασία καρστιά για λόγους χρόνου από κάθε ομάδα που έχει ζητήσει ο μιλητή. Θα δώσω το λόγο σε έναν και μόνο σε εκείνους που δεν έλαβαν το λόγο την τελευταία ώρα. Ο κύριος Πόλτσακ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, για να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι θα δώσετε το λόγο στο συνάδελφό μου. Σας ευχαριστώ όμως. Θα ήθελα να πω ότι ε, μιλήσαμε ε, για τα 800 χρόνια, για τη χάρτα για τα 800 χρόνια, για την ανθρωπιστική προσέγγιση του κόσμου, για τη χάρτα του ανθρωπισμού που δημιουργήθηκε στην Αγγλία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πολλές εθνικές κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν ε, το γεγονός ότι η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για, τις πρόσφυγες, για τις πρόσφυγες έπρεπε να μειώσει την ανθρωπιστική βοήθεια δραστικά σε ένα βραχή χρονικό διάστημα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε αυτές τις πληροφορίες, πώς ε, συνεργάζονται οι κυβερνήσεις όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως την ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία των ανθρώπων. Θα πρέπει να δούμε πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι. Ο παρακαλώ, για ένα λεπτό. you have to put on the microphone, please. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η μητέρα Τερέζα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ είχε πει ότι όταν σκοτώνουμε ακόμα, αυτούς που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, αυτό απειλεί ακόμα περισσότερο την ειρήνη. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά πριν ψηφίσουμε αυτό το έγγραφο γιατί μέσα στα πλαίσια του ανθρωπισμού ορίζουμε και το θέμα της άμβλωσης. Υπάρχουν παιδιά που ζουν σε αυτό τον πλανήτη που δεν θα είχαν γεννηθεί αν ε, όριζαν την κατάσταση οι πολιτικές αρχές. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα πρώτα τελευταίος μέρος της Επιτροπής, ο κύριος Τηλιανίδης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να συγχαρώ τον, συνάδελ, τον ε, συνάδελφο Γκερέρο Σαλόμ για αυτή την εξαιρετική έκθεση και να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την επικοδομητική συζήτηση για την πολύ σημαντική έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τον επόμενο Μάιο στην Κωνσταντινούπολη έχουμε μία ευκαιρία, αλλά ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία, έτσι ώστε το ανθρωπιστικό σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις καταστάσεις μέσα στα πλαίσια των πολυμερών εταιρικών σχέσεων. Η προπαρασκευαστική διαδικασία έχει προωθηθεί, αλλά υπάρχει κίνδυνος ότι η διάσκεψη θα προσπαθήσει να καλύψει τα πάντα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ε, σημαντικά αποτελέσματα θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εξειδικευμένα ζητήματα τα οποία να συστήσουμε εκ των προτέρων με τους εταίρους. έχετε εκτενώς αντιμετωπίσει το θέμα και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα ουσίας. Πρώτον, σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη διαφορά. Θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα επίσης ένα πιο ε, διαφανές σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας με τους οργανισμούς που θα εργάζονται υποκατάσταση διαφάνειας και χρειάζονται και περισσότεροι πόροι και προβλέψιμη χρηματοδότηση. Όλοι το γνωρίζετε. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, νέες χρηματοδοτήσεις, νέες πηγές πόρων στον αναπτυξιακό τομέα Χαίρομαι διότι η Κρυσταλίνα Γεωργίευα, η Επίτροπος θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά η διάσκεψη θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα συγκεκριμένα. Γι' αυτό θα πρέπει να οικοδομήσουμε καλύτερες εταιρικές ε, σχέσεις. Θα πρέπει οι ε, επιτόπιοι παράγοντες να δράσουν ε, ακαρίαια και αυτό αφορά και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Και θα πρέπει να δείξουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εγχείρημα της Δύσης. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας τους επόμενους μήνες, να συνεργαστούμε δημιουργικά, να είμαστε καινοτόμοι, αλλά να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα ζητήματα, έτσι ώστε να μην απεραντολογούμε. Προσμένω λοιπόν στη συνεχή, συνεχή συνεργασία εν ώψη της Κωνσταντινούπολης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο Ενρικέ κύριε Σαλόμ, ως εισηγητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καθόλου τη συζήτηση επιμείνατε όλοι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Καταρχήν, δεν μπορούμε να λύσουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα της μόνο με ανθρωπιστικό τρόπο θα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάποιες σειράξεις και να πετύχουμε κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Μόνο έτσι θα προλαμβάνουμε τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης με περισσότερους δωρητές, με περισσότερους πόρους και χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική της επικράτεια να εφαρμόζει τις ανθρωπαστικές αρχές τις οποίες θα προωθήσει στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο αν δώσουμε το καλό παράδειγμα, το είπε και το ξαναλέω και εγώ, ε, θα είμαστε πιστικοί ε, στην επόμενη διάσκεψη αυτή. Θα ήθελα να συγχαρώ τις πάνω από 30 μη κυβερνητικέ οργανώσεις που συμμετείχαν στην ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής, τους κοιόδης τον Επίτροπο τον κύριο Στυλιανίδη βεβαίως και την Αντιπρόεδρο την κυρία Γεωργίευα και όπως επίσης το προσωπικό το οποίο συνεργάστηκε μαζί μου σας πω πως προσπάθησα η έκθεση μου να είναι ισορροπημένη, να βρω τη χρυσή τομή μεταξύ των θέσεων των διαφέρων ομάδων και λίγες ώρες πριν ψηφιστεί θα ζητούσα από τις ομάδες οι οποίες έχουν αποφασίσει να μην την στηρίξουν να θεωρήσουν τη θέση αυτή γιατί η διάσκεψη είναι πολύ πιο σημαντική από την έκθεση τη δική μου. Όμως η θέση του Κοινοβουλίου είναι και αυτή σημαντική για εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα που περιμένουν στην Κωνσταντινούπολη να αναλάβουμε δράση, δεσμεύσεις και να αποκριθούμε στην ανάγκη να προστατεύσουμε ζωές και να τους σώσουμε από αναξιοπρεπείς καταστάσεις που συμβαίνουν σε τόσους ανθρώπους, σε τόσα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση, η λάβει χώρα αύριο. Και... Κύριε Μαριά. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να θέσω ένα θέμα επί του κανονισμού. Επειδή η ώρα είναι δέκα και δέκα και έχουμε δύο συζητήσεις, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα ακολουθήσετε το θέμα του Catch the Eye. Διότι είμαι εδώ από τις τρεις η ώρα και με διάφορες αιτιολογήσεις η Προεδρία δεν μου έχει δώσει το λόγο ορισμένες φορές. Θέλω να ξέρω λοιπόν αν θα τηρείτε να δίνετε έναν από κάθε ομάδα ή σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο τρεις συνάδελφοι που μπορεί να είναι της ίδιας ομάδας αν θα δώσετε το λόγο. και αυτό να το ξέρω διότι αν είναι να ακολουθήσετε την τακτική που είχατε προηγουμένως θα το γνωρίζω ώστε να μην συμμετέχω και να αποχωρήσω από την αίθουσα. ευχαριστώ. Κύριε Μαριά, έχουμε ήδη πολύ περιορισμένο χρόνο και με βάση τον προγραμματισμό μας ε, υπολογίζουμε να τελειώσουμε στις 11. Γι' αυτό και αποφασίζω η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ να γίνεται έτσι ώστε να λαμβάνει το λόγο μόνο ο μιλητής από κάθε ομάδα που δεν έχει μιλήσει νωρίτερα. Εάν είσαστε βέβαια ο μόνος από την ομάδα σας θα μιλάτε εσείς, αλλά ε, εάν υπάρχει και άλλος που έχει στήσει το λόγο από την ομάδα σας τότε θα μιλήσει ο άλλος συνάδελφος. Δεν μπορώ δηλαδή να δίνω το λόγο σε κάθε βουλευτή που έχει στήσει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα λάβω το λόγο στην επόμενη διαδικασία Καριστέα, γιατί δεν μπορώ να έχω τα ονόματα αυτή τη στιγμή. Και τώρα έχουμε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Πρώτη ομιλήτρια, κύριε Επίτροπος Μαριάννε Τίσαν, την οποία και καλωσορίζω. Σας παρακαλώ να περιορίσετε στα πέντε λεπτά ή δυνατόν.